Και περάσουμε στην επεξήγηση ψήφου. Ο κύριος Σάμπερ πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω ότι ήμουν μόνο ένας από τους πέντε ευρωβουλευτές που κατεψηφίσαμε το ψήφισμα αυτό. Αυτό όχι γιατί δεν θέλω οικονομική βοήθεια σε αυτούς που υποφέρουν τραγικά από την συγκεκριμένη αυτή κρίση και να τους δοθεί βοήθεια. Σωστό να γίνει αυτό. Το έκανα όμως διότι το ψήφισμα αυτό όπως και σε περισσότερα ψηφίσματα για τη Μέση Ανατολή πάσχει. Είναι λοιπές το ψήφισμα διότι δεν αποκαθιστά τα ορθά και τα μη ορθά της κατάστασης. Γι' αυτό το ψήφισμα αυτό δεν έπρεπε να υπερψηφιστεί. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε όσον αφορά τη Γάζα λόγω της δράσης της ομάδας της Χαμάς που στέλνει ρουκέτες και εμβόβε εναντίον ως επικυρίαρχου κράτους που έχει το δικαίωμα ως οποιοδήποτε επικυρίαρχο κράτος να αντιδράσει και να υπερασπίσει τους πολίτες του και μέχρι ότου καταστεί σαφής η ευθύνη για την κρίση αυτή σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου τα ψηφίσματα τα ίδια δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά. Ήρθε καιρός το Ευρωκοινοβούλιο να πει στην Χαμάς αναγνωρίστε το κράτος του Ισραήλ, διαπραγματευτείτε με το Ισραήλ και οι αντισημιτικές απόψεις βγάλτε τις από τον χάρτη σας. Τότε θα αρχίσει η ειρηνευτική διαδικασία. Πρόεδρος. Περνάμε στην έκθεση Κίνοκ. Η κυρία Τομασιούσκα. Κυρία Πρόεδρε, είναι απαραίτητη η ανάληψη ευθυνών από τους γονείς και τους ενήλικους για την ζωή των παιδιών. Γιατί πολλές φορές αναμειγνύονται και σε έναπλες συγκρούσεις, εκτίθεται στη, στο θάνατο, στην έλλειψη φαρμάκων, στον υποσυτισμό. Εγώ παρόλα αυτά καταψήφισα την έκθεση αυτή γιατί τάσεται υπέρ των αμβλώσεων. Αυτό πραγματικά είναι παράλογο. Πώς είναι δυνατόν να ισχυριζόμαστε ότι προσπίζουμε τα συμφέροντα των παιδιών ενώ δεν υπερασπιζόμαστε καν το δικαίωμα στη ζωή. Ευχαριστώ κυρία Σίνοτ. Oh, Ο κύριος Καμάλ. Κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Δείξτε τους την ομορφιά που έχουν μέσα τους, είπε η φιλόσοφος Χούιτνη Χιούστον. Για πρώτη φορά με την έκθεση αυτή εξετάζουμε πραγματικά το κλειδί για τη, για μελλοντική ανάπτυξη. Και αυτό που είναι σημαντικό επίσης είναι ότι εξετάζουμε την ανάπτυξη των παιδιών και την διαπαιδαγωγησή τους και όχι μόνο των κοριτσιών γιατί εκπαιδεύοντας τα κορίτσια εκπαιδεύεται και μια μελλοντική γυναίκα και επομένω μια μελλοντική μητέρα και μια ολόκληρη οικογένεια. Ζητώ από όλους τους συναδέλφους μας να εξετάσουν τις λύσεις που ε, προτείνει το Πανεπιστήμιο του Newcastle και θεωρεί ότι όπου το κράτος δεν έχει προσφέρει επαρκή διαπαιδαγώγηση στα παιδιά έχουν φροντίσει οι γονείς συνερχόμενοι σε οργανώσεις και ζητώ να τους υποστηρίξουμε. Η κυρία Εγώ καταψήφισα την έκθεση εκείνο με βαριά καρδιά γιατί τα προβλήματα που εντοπίζει είναι πολύ σημαντικά. Τραγωδίες συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο αλλά η βάση της εκθέσεώς της είναι η Σύμβαση των ΗΠΑ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και προχωρούμε στη βάση μιας πολύ ελληματικής ε, συνθήκης. Πάντοτε είχε προβλήματα η συνθήκη αυτή. Αφενός περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία, από την άλλη πλευρά περιλαμβάνει και ορισμένα εντελώς ακατάλληλα ε, σημεία. Γράφτηκε το 1989. Έχει, για παράδειγμα, περιλαμβάνει για παράδειγμα ε, το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για τα παιδιά και υπέρ των παιδιών πριν να γνωρίζουμε τα σχετικά με αυτούς που καταχωρώνται τα παιδιά μέσω ε, των ε, μέσων ενημέρωσης. Και βάζει και το κράτος ως μοναδικό διαιτητή που και κριτή του βέλτου συμφέροντος του παιδιού. Ξεχνώντας τους γονείς ή τα νηπιαγωγεία ή τους άλλους που τα φροντίζουν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκα να καταψηφίσω. Και βάζει και την άμβλωση μέσα, η οποία δεν έχει απολύτως καμία δουλειά μέσα σε ένα κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών. Ένα λεπτό παρακαλώ για τις αιτιολογήσεις ψήφου. Χάνουν. Ευχαριστώ. Οι ψηφοφόροι μας θα ενδιαφερθούν να μάθουν πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει στους ε, τομείς αυτούς. Πριν από το Ιρλανδικό Δημοψήφισμα και μετά μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρεί σε κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε πρόκειται να ανακατευτεί σε θέματα νόμων αμβλώσεων. Να όμως που τώρα συγχωνεύονται τα δύο αυτά θέματα σε μια έκθεση. Όλες οι υποσχέσεις λοιπόν που έχουμε δώσει ότι θα ακούμε τι λένε οι άνθρωποι και ότι θα ράβουμε και θα κόβουμε τις ε, πολιτικές μας για να τους βολεύουν, ήταν άχρηστες. Τα ακούσαμε και ακούσαμε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίο εκφώνησε ε, λόγο ε, πλήρη ε, κοινών τόπων. Και εν τέλει, ποια ήταν η αντίδραση ε, του Κοινοβουλίου όταν είπε ότι πρέπει να ακούμε και τους άλλους, τις άλλες απόψεις. Βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και, της, ε, και των Σοσιαλιστών σηκώθηκαν και βγήκαν από την αίθουσα. Δεν μπορούν καν να ακούσουν τις απόψεις των άλλων. Εάν λοιπόν νομίζετε ότι κάνω λάθος, τότε να αποδείξετε ότι κάνω λάθο, να διεξαγάγετε τα δημοψηφίσματα που ήδη ούτως ή άλλως έχετε υποσχεθεί. Κυρία Τομασέφσκα, για την έκθεση Κοτινή. Κυρία Πρόεδρε, η μετάθεση της οδηγίας 2002-2030 για την ε, διαβούλευση με τους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα την εποχή της κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κάποιες δεσμεύσεις που έχουν σχέση με την κοινωνική ευθύνη. Ε, όταν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την, ε, την, την, όταν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την απασχόληση ή την εκπαίδευση των εργαζομένων. Η μετάθεση της οδηγίας θα πρέπει να επιταχυνθεί στις χώρες μέλη και να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση Κοτίνη. Ευχαριστώ. Έκθεση Τόγεν η επόμενη. Ο κύριος Σεκέρσκι. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται υπέρ τη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και η στρατηγική τη Λισαβόνα ε, θέλει να προωθήσει και τι θέσει απασχόληση. Επίση, ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε την ανάγκη προστασίας της υπαίθρου ε, και την προστασία των βιομηχανικών ζωνών και των βιομηχανιών γενικά που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά χρειάζονται για τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη και την επίλυση των νέων οικονομικών προβλημάτων. Βέβαια, ορισμένες παραδοσιακές βιομηχανίες θα πρέπει επίσης να προστατευτούν θα πρέπει να τονώσουμε την βιομηχανική ανάπτυξη, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε και την κοινωνική ανάπτυξη. Η κυρία Τομασέφσκα και πάλι. Κυρία Πρόεδρε, η χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε προβλήματα ακόμη και στην ε, ελεύθερη διακίνηση των πολιτών που έχει και κοινωνικές αλλά και οικονομικές ε, επιπτώσεις όπως η συμμετοχή στο Ε.Π. Κάθε νέα θέση απασχόλησης, κάθε νέα ποιότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες έχει πια τη δική της αξίας. Είμαι υπέρ της έκθεσης και περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα προσέγγιση και οργανωτική και χρηματοπιστωτική τονίζοντας την κοινωνική οικονομία, ιδιαίτερα μέσω της απλούστευσης των διοικητικών μηχανισμών με τη χρησιμοποίηση κοινοτικών κονδύλιων. Γι' αυτό, όπως σας είπα, υπερψήφισε την έκθεση. Ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Διαβάζοντας την έκθεση αυτή είδα τον ορισμό της κοινωνικής οικονομίας και με ενδιαφέρουν κοίταξα τι λέει αυτός ο ορισμός και λέει δύο ταξίς που παραξένευσαν Τώρα οι κοινωνικοί στόχοι έναν του κεφαλαίου και άλλη της εγκληγής και ευθύνης και δημοκρατικός έλεγχος από κράτη-μέλη. Δεν αναφέρεται καθόλου η ελεύθερη προαιρετική ανταλλαγή μεταξύ παραγωγού και αγοραστή που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα ήταν πιο κοινωνικό από το να κάνει κανείς ένα όφελος, να ξαναεπενδύσει, να δημιουργήσει απασχόληση για το καλό όλων. Όταν αρχίζουμε να κοιτάμε τις κοινωνικές ανάγκες και όχι την ίδια την ανάγκη του να δημιουργηθεί και κέρδος που θα οδηγήσει στη δημιουργία απασχόληση και στη διασπορά του πλούτου στην κοινότητα, πέφτουμε στην παγίδα που μας προειδοποίησε ο Αυστριακός οικονομολόγος στις αρχές του αιώνα και άλλοι οικονομολόγοι όταν ξεχνάει κανείς το κέρδος κινούμαστε στον κατηφορικό δρόμο της δουλείας και γι' αυτό καταψήφισα αυτή την έκθεση. Πρόεδρος. Έκθεση Τζαμπάζη για την ψυχική υγεία. Κυρία Ντόιλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρά την ψυχική υγεία και τη αποδίδουμε προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντική στο πρόγραμμα Υγεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γιατί μέχρι το 2020 οι ψυχικέ ενώσει θα είναι από τι πιο σημαντικέ στον αναπτυσσόμενο κόσμο και στη δική μου πατρίδα έχουμε την θεωρία περισσότερο να μιλούμε και λιγότερο να έχουμε αυτά έργα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τώρα την προσέγγιση μας και πολλές ε, δράσεις της έκθεσης ε, ε, περιορίζονται στην εθνική πολιτική αλλά και περιχαρακώνται πολλές φορές από την ευρωπαϊκή πολιτική. Δυστυχώς όμως ε, υπάρχει τεράστια αποσύνδεση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης, των καλών λόγων, των εκθέσεων και των δράσεών μας. Έχουμε προγράμματα δράση που αποφεύγουν τη δράση. Θα πρέπει πραγματικά να λάβουμε σοβαρά υπόψη την ψυχική υγεία που είναι η σταχτοπούτα δυστυχώ των πολιτικών ψυχική υγεία των ε, χωρών μελών. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Η κυρία Νίνα Γκίλ, ένα στου τέσσερι ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας τουλάχιστον μία φορά στο βίο τους. 8 από τις δέκα βασικές αιτίες ε, της ανικανότητας είναι θέματα ψυχικής υγείας και τα ψυχικά προβλήματα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα θύματα αυτών των νόσων. Θα πρέπει λοιπόν να εξυγχρονίσουμε την ε, νομοθεσία περί ψυχικής υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτής της ψυχικής υγείας. Θα πρέπει ε, να πούμε στους ψηφοφόρους ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, τα σχολεία, όλα, όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες για την ψυχική υγεία και διασύνδεση μεταξύ των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας και ε, εξήγηση ε, και πρόταση να να, χρηματοδοτούν η να χρηματοδοτηθεί η ψυχική υγεία από το Περιφερειακό Ταμείο και τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Επίση, θα δούμε το στρες που σχετίζεται με την εργασία, το εργασιακό περιβάλλον, να αντιμετωπίσουμε τι στρεσογόνους παράγοντες στην εργασία. Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να ε, προωθηθούν. Σα ευχαριστώ κύριε Γκίλη. Κυρία Τομασεύσκα. Κυρία Πρόεδρε. 90% των αυτοκτονιών οφείλονται σε ψυχικά προβλήματα και αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από κατάθλιψη ή άλλες ασθένειες του πολιτισμού εξαιτίας του στρες που υφίστανται και του ρυθμού της ζωής τους. Στην ε, Ευρώπη έχουμε όλο και περισσότερο ψυχασθενείς και μάλιστα σε νωρίτερη ηλικία η αποφυγή της, της διάγνωσης της ψυχικής υγείας, ο στιγματισμός μερικές φορές, η υποστήριξη της οικογένειας ε, δεν ε, γίνεται σωστά. Όλα αυτά όμως ε, επηρεάζουν την κοινωνία και αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε άμεσα δράση. Είμαι υπέρ της έκθεσης κυρία Τζαμπάζη και την υπερψήφισα. Η κυρία Σίνοτ. Και εγώ υπερψήφισα τη έκθεση, αλλά χάσαμε μια ευκαιρία κατά τη γνώμη μου έπρεπε να συμπεριλάβουμε και τα ηλεκτροσόκ. Δηλαδή να προτείνουμε ολοσχερή απαγόρευση αυτού, αυτής της βασανιστικής μορφής θεραπείας που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε πολλές ε, ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ε, τάση να εξετάζονται παιδιά για ψυχικά προβλήματα και σωστή σωστή φαρμακευτική αγωγή. Δυστυχώς δεν είναι αρκετά φιλόδοξη η έκθεση από αυτή την άποψη. Ε, αναφέρεται το θέμα της εξέτασης των παιδιών. Γιατί δεν φαίνεται φυσιολογική η η εξέταση από πολύ παιδική ηλικία. Πάντως, δεδομένη τις έξαρση αυτών των προβλημάτων ψυχικής υγείας, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αίτια αυτής της έξαρση, ιδιαίτερα για τη αυτοκτονίας. Φαίνεται ότι η κοινωνία μας δεν επιτρέπει τον υγιή τρόπο ζωής. Γιατί αν επιδεινώνεται η ψυχική υγεία θα πρέπει να δούμε τι κοινωνία διαμορφώνουμε. Ευχαριστώ. Περάμε στην έκθεση Γκιούρκ. Ο κύριος Ρουτόβιτς. Κυρία Πρόεδρε, είμαι κατά της έκθεσης και του ψηφίσματος και καταψήφισα για τους εξής λόγους σοβή χρηματοπιστωτική κρίση και τα θεσμικά όργανα έχουν σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Οι δαπάνες της Ένωσης ε, είναι υπερβολικές και πολλές φορές ε, έχουμε αθώα θύματα τέτοιων ε, δράσεων εγκληματικών. Δεν μπορούμε λοιπόν με τα σχέδια αυτά να ενισχύουμε ουσιαστικά τους παρανόμους. Επίσης, μερικές φορές ε, για λόγους ψηφοθυρίας ε, περιοριζόμαστε στα λόγια και δεν αξιοποιούμε σωστά τα κονδύλια της Ένωσης και τα, την προσφορά των φορολογουμένων. Στο μέλλον, όταν έχουμε παρόμοια προβλήματα, θα πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Έκθεση Ράμος. Κυρία Ντόιλ έχει εξήγηση Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επικροτώ ιδιαίτερα την έκθεση της κυρίας Μιγγέ Δράμος για την εφαρμοσμένη έρευνα στο τομέα της κοινής αλληλευτικής πολιτικής για να εφαρμοστεί η εφαρμοσμένη έρευνα. Η προστάτευση του ε, αλληλευτικού πλούτου είναι αναγκαία προκειμένου να πετύχουμε μια σωστή, σωστή ισορροπία χρησιμοποιώντα την πιο προφημένη και επίκαιρη επιστημονική τεχνολογία θα μας βοηθήσει. Ωστόσο, θα ήθελα να προσέξουμε κάτι. Στους δύσκολους οικονομικούς χειρούς που περνάμε, πρέπει να φυλαγόμαστε από επικάλυψη προσπαθειών, να την αποφεύγουμε. Πρέπει να φροντίσουμε σε κοινωτικό επίπεδο να μην κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κεμάλ. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για εφαρμοσμένη έρευνα, πρέπει να δούμε και τα ατελή σημεία της αλληλευτικής πολιτικής. Έχουμε κοινή αλληλευτική πολιτική εδώ και 40 χρόνια με στόχο να έχουμε βιωσιμότητα του κλάδου. Αλλά δεν το πέτυχε αυτό, ούτε καν η προστασία του περιβάλλοντος. Έπειτα έχουμε τα ε, δικαιώματα που έχουν χώρε, όπω η Νέα Ζηλανδία που διαπίστωσαν ότι δίνοντα, προστατεύοντα τα συμφέροντα αυτό που εργάζονται στον κλάδο, το πετυχαίνουν καλύτερα. Μια προσέγγιση δηλαδή που να στηρίζεται περισσότερο στην αγορά με ε, ανταλλαγή ατομικών ποσοστώσεων. Φυσικά μπορούμε να εφαρμόσουμε τη νέα έρευνα, τη νέα τεχνολογία, αλλά αν εξακολουθήσουμε να κρατάμε ένα σύστημα παρόλες τις καινοτομίες όπου οι κυβερνήσεις λένε στον κάθε αγία πόσο θα πρέπει να αλλιεύσει, όλη η εφαρμοσμένη έρευνα θα είναι χαμένος χρόνος. Είναι καιρός να καταργήσουμε την κοινή αλλιευτική πολιτική. Ας προχωρήσουμε στην έκθεση Βάντενμπεργκ. Έγια Μακκίλ. Στα πλαίσια αυτή της ε, δύσκολης οικονομικής συγκυρία, προσφέρει ιδέες που είναι απαραίτητε η παρούσα έκθεση. Οι μειώσεις αυτές ε, θα επιτρέψουν σε πολλούς να αναπνεύσουν. Επίσης η έκθεση αναφέρεται στην προσπάθεια δημιουργία απασχόλησης και αυτό την υποστήριξα. υποστήριξα. Ελπίζω ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα που προτείνει γρήγορα και ιδίω στην περιοχή μου, στα West Midlands. Τονίζω επίσης ότι πρέπει οι χώρε μέλη να έχουν το δικαίωμα να μειώσουν τους συντελεστέ ΦΠΑ σε ορισμένου τομείς για να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανάγκες προστασίας του κλίματος, ώστε να υπάρξουν και κίνητρα υπέρ τη αγορά πράσινων προϊόντων, οικολογικά ασφαλών προϊόντων. Οι μειώσει του ΦΠΑ χρησιμοποιούνται παντού ως κίνητρα για τους καταναλωτές για να αγοράσουν περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα όπως σύγχρονες τεχνολογίες, ψυγεία κλπ. Η κυβέρνησή μου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει πρωτοπόρο ρόλο μειώνοντας κατά 2,5% τον ΦΠΑ μέχρι το 2010. Ελπίζω και άλλες χώρες να πράξουν όμοια. Ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ. Κύριε Πρόεδρε, η μόνη μάχη που σίγουρα θα χάσουμε είναι αυτή που δεν θα ξεκινήσουμε με την επανυποβολή των τροπολογιών για ε, πιο δίκαιη εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ιδιαίτερα για τα παιδικά ενδύματα στις νέες χώρες μέλη. Αποκαθιστούμε την ίση μεταχείριση με τις παλιές χώρες μέλη και θέλουμε να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι τα καταφέραμε με μία εξαίρεση να ε, κερδίσουμε τις τροπολογίες μας ε, με εξαίρεση τα εστιατόρια ε, και μάλιστα παρατρίχα θα χάναμε την τροπολογία μας για νέο συντελεστή στα εστιατόρια και όχι δύο διαφορετικούς συντελεστές ε, για τα τρόφιμα και τα ποτά όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το κείμενο προτείνει διαφορετικούς ε, συντελεστές ανάλογα με τις ε, υπηρεσίες των εστιατορίων. Άλλος συντελεστής ισχύει για τα τρόφιμα και άλλος για τα εινοπνευματόδια. Δεν νομίζω ότι κατάλαβαν πολλοί συνάδελφοι την έννοια της τροπολογίας μας. Πάντως το μήνυμα του Κοινοβουλίου και στον τομέα αυτό ε, ισχύει και πραγματικά άξιζε, άξιζε αυτή η μάχη που δώσαμε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που επιμείναμε στην ομάδα μας για να καταπολεμήσουμε αυτή την κακή μανία της ε, ε, δημευτικής φορολογίας της αριστεράς. Θα πρέπει να, να πατάξουμε αυτή την φορολογομανία Σάμπερκ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ίσως πρόκειται για το δυσχερέστερο θέμα για μια ελεύθερη κοινωνία. Πώς αντιμετωπίζει μια ελεύθερη κοινωνία εκείνους που επιθυμούν να την καταστρέψουν. Και αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία και βέβαια πρέπει να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ασφαλώ και πρέπει να σεβόμαστε τι νομικέ διαδικασίε. Ορισμένε φορέ όμω, στον κόσμο που ζούμε σήμερα, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Στην Ευρώπη και στις χώρες της Ευρώπης δεν μπορούμε να επαφιέμεθα μόνο στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην χώρα μου δικάζονται αυτή τη στιγμή οκτώ άτομα τα οποία ε, κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να αναδυνάξουν στον αέρα οκτώ αεροπλάνα. Δεν τα κατάφεραν ευτυχώς. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι η ελεύθερη κοινωνία θα έχει τους μηχανισμούς και τα μέσα για να νικήσει εκείνους που προσπαθούν να την καταστρέψουν. Εάν δεν το επιτύχουμε αυτό, τότε αποτυγχάνουμε στην προσπάθειά μας να υπερασπίσουμε αυτούς που μας στέλνουν εδώ. Ρούτοβιτς. Συγγνώμη, είχα ήδη μιλήσει για το θέμα αυτό. Ε, σας ευχαριστώ. Έκθεση Φων Βόγκαου, κ. Μπέργκ. Εγώ ζήτησα και από τους άλλους Ιρλανδούς βουλευτές να απόσχουν από την ψηφοφορία της έκθεσης ε, Βόγκαου αλλά και Βάτανεν διότι η Ιρλανδία έχει διατηρήσει την ουδετερότητά της και στο σχετικό πρωτόκολλο εγγράφεται αυτό. Έχει ένα τριπλό σύστημα προστασίας η Ιρλανδία. Χρειάζεται δηλαδή εντολή των Ηνωμένων Εθνών, έγκριση από την κυβέρνηση και έγκριση από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο για να συμμετάσχουν οι Ιρλανδικέ δυνάμει σε οποιαδήποτε εξωτερική αποστολή. Και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και υπό την Λισαβόνα. Δεν σημαίνει ότι η Ιρλανδία δεν θέλει να παίξει το ρόλο τη. Ιδιαίτερα σε ειρηνευτικέ αποστολέ συμμετέχουμε, για παράδειγμα στο Τσάντ, με ιδιαίτερα επιτυχή τρόπο. Με εντολή των Ηνωμένων Εθνών, όπου τα Ηνωμένα Έθνη δεν είχαν επαρκή δυνάμει και παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει. Η εντολή αυτή λήγει 15 Μαρτίου. Ωστόσο πέρασαν 18 μήνες ιδιαίτερα επιτυχούς προσπάθειας και θα συνεχίσει η προσπάθεια αυτή και η Ιρλανδία θα συνεχίσει να συμβάλλει σε ειρηνευτικές αποστολές είτε των ΗΕ είτε της Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ. Έκθεση Κύριε Κέλαμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την παράγραφο 43 της εκθέσεως Βατάνεν μόνον επειδή υπέβαλε προφορικές τροπολογίες ο κύριος Λαντσμπέργκης. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει καλύτερα η αρχική παράγραφο 43 που λέει ότι οι προτάσεις ασφαλείας που έχει καταθέσει πρόσφατα η Ρωσική Κοινοπολιτεία υπονομεύουν την αξιοπιστία των ε, δομών ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, ε, βάζουν προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχοντας παρακολουθήσει τις εργασίες της ε, Επιτροπής Συνεργασίας Ενώσεως Ρωσίας, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια πραγματικότητα που είναι ότι η Ρωσία προσπαθεί να βάλει μια σφίνα ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους και στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Σόμπερκ, ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σχολιάσω σύντομα αυτό το θέμα. Ήταν αξιοθαύμαστη ομιλία του Τσέχου Προέδρου που μας υπενθύμησε την ιστορία της πατρίδας του αλλά και άλλων χωρών, ιδιαίτερα της Ανατολικής Ευρώπης, που υπέστησαν την ναζιστική κατοχή αλλά και την ε, επόμενη κομμουνιστική κατοχή. Αυτό δείχνει τη ζωτική σημασία που έχει το ΝΑΤΟ και η διατήρηση του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει στην κοινωνία. Αλλά η βασική πρωταρχική άμυνα του, της Δύσης θα εξασφαλιστεί από το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η συμμαχία μας με, τους, ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και κάτι ενοχλητικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που το διαπιστώνουμε πολλές φορές, είναι μία λαθάνουσα και μερικές φορές φανερή τάση αντιαμερικανισμού. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν αυτές που μας επέτρεψαν να μιλούμε σήμερα ελεύθερα και το ΝΑΤΟ εγγυάται αυτή την ζωτική συμμαχία και για το μέλλον. Ο κύριος Καμάλ και πάλι. Σας ευχαριστώ. Στο μεγαλύτερο τμήμα του προηγούμενου αιώνα και μέχρι στιγμή στο δικό μα αιώνα, το ΝΑΤΟ συνέβαλε στη διατήρηση τη ειρήνη. Υπάρχουν όμω κάποιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλουν να υπονομεύσουν το θεσμό αυτό, το θεσμό που μα επέτρεψε να συνεργαστούμε με του ε, Αμερικανού και Καναδού συναδέλφου και πολλέ ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούν να υπονομεύσουν το ΝΑΤΟ, όχι μόνο με άμεση επίθεση προ το ΝΑΤΟ, αλλά με αλληλεπικάλυψη των δομών του. Φαίνεται ότι έχουμε μια κατάσταση που Αμερικανοί και Καναδοί ε, συνέρχονται με, Αμερικανούς, ε, με Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες ε, υπό την ηγέτα του ΝΑΤΟ και η ίδια συνεδρίαση θα γίνεται αλλά χωρίς τους Καναδούς και τους Αμερικανούς μια επανάληψη ουσιαστικά της ίδιας συνεδρίασης. Αυτό είναι διασπάθηση χρόνου και πόρων. Είναι ζωτικό ο ρόλο του ΝΑΤΟ και α μην ξεχνούμε, ένα τμήμα του ΝΑΤΟ είναι ο καταμερισμό του βάρου. Και αν έχουμε ε, μηχανισμό άμυνας, μόνο η Γαλλία και η Αγγλία θα μοιραστούν αυτό το βάρος, ενώ οι άλλοι θα μείνουν πίσω. Ας μην ξεχάσουμε το σωτικό ρόλο που έπαιξε το ΝΑΤΟ και θα πρέπει να συνεχιστεί. Ο κύριο Μπέρκ. Θα ήθελα να προσθέσω αυτά που είπα προηγουμένω ότι περιμένουμε να κυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας ε, από την Ιρλανδία, αλλά θέλουμε να διαφυλάξουμε την ουδετερότητά μας και με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεν θα υπαναχωρήσουμε ως προς αυτό. Θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε το ρόλο μας, αλλά με φιλιρινικό τρόπο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και στο παρελθόν συμμετείχαμε σε ε, επιχειρήσεις διατήρησης της και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Ο κύριος Μοντάλτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους υπαλλήλους. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 17 που ήταν μετά τη 45, έπρεπε να ψηφιστεί μετά τη 45 και εγώ και ο κύριος Γκρέκο, παρακαθήμενος θέλαμε να ταχθούμε υπέρ της αποστρατικοποίησης του διαστήματος. Εκείνη όμως τη στιγμή της ψηφοφορίας αποσπάστηκε η προσοχή μας από κάποιο γεγονός και δυστυχώς από αφηρημάδα δεν μπορέσαμε να το ψηφίσουμε. Καλώς. Περνάμε στην έκθεση Ναπολετάνο. Ο κύριος Μουσουμέτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 14 χρόνια από τη διάσκεψη της την μεσογειακή εταιρική σχέση, ο απολογισμός είναι τελείως μη ικανοποιητικός σε σχέση με τις ε, οικονομικές δεσμεύσεις είναι κάτι θεμητό να το κάνει το Κοινοβούλιο και υποχρέωση της Κομισιόν να αποδώσει λογαριασμό. Τα ατομικά δικαιώματα δεν προστατεύονται απόλυτα σε όλη αυτή τη ζώνη σε σχέση με τη θρησκευτική ελευθερία δεν υπάρχει ακόμη μια πλήρη ευχή η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ακόμα είναι στο σημειωτόν ενώ το ανθρωποεμπόριο που τροφοδοτεί τους παράνομους μετανάστες ιδιαίτερα στις, ακτές της χώρας μου Νότια Ιταλία, Σικελία με όλα αυτά τα δεδομένα να ανοίξει μια ελεύθερη ζώνη δεν είναι ευκαιρία, αντίθετα αυξάνει την απόκληση και το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών περιοχών. Ιδιά με τις παραγράφους 29 και 36 αυτή την επιφύλαξη η ομάδα μου ψήφισε υπέρ της διαδικασίας Βαρκελόνης ως μια χειρονομία ελπίδας, παρότι έχουμε όλους αυτούς τους δισταγμούς. Προχωρούμε στην έκθεση Σιμάνσκι. Ο κύριος Σικιάρσκι. Ευχαριστώ πολύ. Η εταιρική σχέση με την Ανατολή είναι σημαντική και θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα της πολιτικής γειτονίας της Ένωσης. Θα αναφερθώ σε τέσσερα σημεία κλειδιά Πρώτον, πρόθεση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα στις χώρες αυτές και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, οικονομική ολοκλήρωση. Θα πρέπει να μπορέσουν όλοι να έχουν πρόσβαση σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου τους και προάσπιση των δικαιωμάτων τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση κρίσης. Διασφάλιση της σταθερότητας ε, της Ευρώπης και της ενεργειακής της ασφάλειας. Θα πρέπει να αποφευθούν κρίσης ε, φυσικού αερίου εξαιτία του μονοπωλίου των προμηθευτών ε, ή των ε, μέσων μεταφοράς. Επίσης θα πρέπει να τονώσουμε τις πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές. Έτσι θα βελτιώσουμε το προφίλ της Ένωσης προς Ανατολάς και θα δώσουμε παράδειγμα ανοχής και συνεργασίας η ανατολική γειτονία χρήζει ιδιαίτερης και προσεκτικής συζήτησης. Και τέλος, έκθεση Ντόλ, ο κύριος Κορμπέτ, για δύο λεπτά από την ομάδα του. Με ιδιαίτερη χαρά υπερψήφισα την έκθεση και εύχομαι ε, καλή αδιαμητρότητα στην κυρία Ντάλ. Ως μέλος της ε, Ομάδα της ε, ζήτησε να αναλάβει αυτή την έκθεση προκειμένου να συμβάλλει και αυτή επικοδομητικά στο έργο του Κοινοβουλίου σε αντίθεση με τους συναδέλφους της από το κόμμα της ανεξαρτησία που ποτέ δεν ανέλαβαν εκθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Το μόνο που κάνουν είναι ε, εξαιτία τη της άγνοιάς τους ε, να κάνουν κάποιες σποραδικές επιθέσεις προκειμένου ε, να εξασφαλίζεται τάχα καλύτερος έλεγχος ε, της ε, κοινοτικής νομοθεσίας και να εκπροσωπούνται τα διάφορα συμφέροντα. Το μόνο που θέλουν όμως οι συνάδελφοι αυτοί είναι να είναι αρνητικοί και να δείξουν πλέον αντιλογία σε όλα. Πού έγκυται το επικοδομητικό της συμπεριφορά τους. Έχω λάβει από το Συμβούλιο τέσσερις κοινέ θέσεις και τους λόγους για την ε, υιοθέτησή τους, καθώς και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τίτλοι θα περιληφθούν στα πρακτικά της παρούσας συνόδου και το τρίμηνο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στη θέση του θα αρχίσει να τρέχει από αύριο 20 Φεβρουαρίου του 2009. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο για έγκριση